Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε, να μην καθυστερήσουμε, γιατί έχουμε και ψηφοφορίες. Καθίστε. Στο σημείο 1, έγκριση της ημέρης της Η ψηφοφορία για το κείμενο που συμφωνήθηκε για τη νομική αρρωγή προς τους υπόπτους ή κατηγορούμενους και σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό δελμά ο κύριος Ντένις Τεγιόμ, ο εισηγητής, ε, θα πάρει το λόγο πριν από το σημείο 3. Αν λοιπόν δεν έχει συντηρήσει στην τροποποιημένη ατζέντα, εγκρίνεται σε ό,τι αφορά την ε, διερμηνία. Τσέχικα, Μαλτέζικα, Λιθουανικά, Δανέζικα και άλλες γλώσσες δεν υπάρχει δυστυχώς σήμερα. Ελληνικά μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε πάντως. Αν είστε έτοιμοι λοιπόν συνάδελφοι, διαδικαστικό να πω ότι ξέχασα την ε, κάρτα μου στην Ολομέλεια και εγώ, λέει η κυρία Σίπελ. Okay. Okay, colleagues, I want... Συνάδελφοι, να μην καθυστερούμε. Ούτε σας παρακαλώ καθίστε. Δύο μέλη δεν έχουν κάρτες μαζί. Δεν προλαβαίνετε να πάρτε να τις πάρετε. Θα σας ε, καταμετρήσουμε όμως. Μήπως κανείς άλλος έχει ξεχάσει την κάρτα του. Να το πείτε τώρα θέλετε. Όχι. Πολύ ωραία. Έχουμε δύο μέλη των σοσιαλιστών και δημοκρατών που δεν έχουν τις κάρτες τους. Θα σηκώνουν το χέρι. Καθίστε παρακαλώ όλοι σας. Okay.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 Έχουν όλοι κάτσει. Άξελ, παρακαλώ, κάτσε. Μάριο, έχει την κάρτα σου, ναι, ναι, ναι. Έτοιμοι Ωραία. Έχουμε μένα τρει συναδέλφου χωρί την ε, κάρτα. Αυτοί πρόκειται να εκφράζονται με ανάταση τη χειρό. Τρει, τρει. Άλλο πριν ξεκινήσουμε, ωραία φύγαμε. Τώρα έχουμε ε, δικαστική συνδρομή για ε, υπόπτους ε, και σε σχέση με το, το ευρωπαϊκό ένταλμα. Ο κύριος Ντεγιόγκ είναι ο συγκητής και αν δεν θέλει το λόγο συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Στην πρώτη ολομέλεια του θα γίνει η ψηφοφορία στον Λομέλη. Τι έχετε διαδικαστικό. Ψηφίζουμε. Just, just raise your hand. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Colleagues, there is one too many... Uh... Ένας παραπάνω, συνάδελφε. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Okay, and now the vote is closed. Πέρασε ο εγκρίνεται. 44-1. Καμία εποχή και συγχαρητήρια εισηγητά. 1η Οκτωβρίου στην ε, Ολομέλη. Θέλετε κάποιο σύντομο σχόλιο. Όχι, καλώς. Κύριε Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι, θέλω να ευχαριστήσω τους χιόδους εισηγητές γιατί ε, τώρα αυτούς τους τελευταίους μήνες δουλέψαμε εντατικά και επιταχύναμε τους ρυθμούς μας κατά την Ελληνική Προεδρία ε, είχαμε την αρχική θέση του Κοινοβουλίου που δεν μπορέσαμε να προωθήσουμε τις θέσεις μας σε σχέση με την ε, οδηγία για διορισμό συνηγόρου Τελικά πάντως για, για την δέσμοι των ε, διατάξεων που εγκρίθηκαν δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγιόγκλη ο και τώρα προχωράμε στο σημείο υπαριθμών 3. Δηλαδή κατάρτιση κοινού καταλόγου των ε, ασφαλών ε, χωρών για την διεθνή συνεργασία. Κυρία Σεβικηγιόμ είναι η συγκίτρια. Τώρα θα εγκρίνουμε το σχέδιο κειμένου και θα ψηφίσουμε επίσης την έναρξη των διαπραγματεύσεων και τη σύνθεση της ε, διαπραγματευτικής ομάδας. Εδώ έχουμε διάφορες ε, διατάξεις που έχουν εγκριθεί και επίσης θα σας πω ότι το 35, το το 108, το 109 και το 119 ε, έχουν αποσυρθεί. Και το 103 μου είπαν σήμερα το πρωί. Οπότε για πέστε μου τώρα, κυρία Σιγήτρια, θέλετε μήπως το λόγο. Όχι. Οπότε τώρα θα ψηφίσουμε. Ξεκινούμε με το 30. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφορίας. Πάλι ένας παραπάνω από το έλεγχο. Πέρα ψηφορίας. Πέρα ψηφορίας. Πάλι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται. 31. Συμβεστική 1. Ψηφίζουμε. Πέρας της πληροφορίες. Εγκρίνεται. 76. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 77. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 9. Τι άφετ. Ψηφίζουμε. Α, συγγνώμη συνάδελφοι, πάμε στο συμβαστικό 2 ψηφίζουμε. ψηφορίες. Εγκρίνεται. Εννέα της ΑΦΕΤ τώρα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τρία ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Ψηφίζουμε. Συμβαστική 5. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφορίες. Και εγκρίνεται. 7. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφορίες. Και εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 104. Ψηφίζουμε. Το 103 έχει αποσυρθεί. Επομένως ε, ψηφίζουμε για το 104. Πέρα ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της συμβαστική 9. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται Συμβαστική 10. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 110. Ψηφίζουμε. Τι θέλετε το αποτέλεσμα, δεν, δεν το είδατε. Για τη 10. Στο τέλος, στο τέλος. Να σας πούμε ακριβώς. Είμαστε τώρα στο 110. Ψηφίζουμε. Τώρα. 110. Τώρα ψηφίζουμε. Πέρασε και εγκρίνεται. 11, συμβαστική 11, ψηφίζουμε. Πέρας και εγκρίνεται. Εκατόν τέσσερα. Ψηφίζουμε το 114. Πέρας. Απορρίπτεται. 115. Πέρας ψηφορίας. 116 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Και απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 120 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. 121 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. 122 ψηφίζουμε. Πέρασε. Και απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 ψηφίζουμε. Και πέρασε ψηφορίας. Και εγκρίνεται. 14 συμβιβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τις ιδεολογικές παραγράφους. Πρώτη. Εγκρίνεται. Παριθμών 2 και 36 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρασε. εγκρίνεται. Σαράντα ψηφίζουμε. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Ψηφίζουν. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 51. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 52. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική. Όχι διορθώνει ο πρόεδρο Πέμπτη αιτιολογική και είναι ταυτόσιμε οι 58 Πέρας. Δεκτή. Τοπολογία 1 της ΑΦΕΤ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 17 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2 της ΑΦΕΤ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 68. έρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Εβδομήντα ένα άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, πλησιάζουμε. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Δεκτή. Το κείμενο όπως τροποποιήθηκε, να έρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Δεκτή, 36 υπέρ, 10 κατά 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Τώρα, συνάδελφοι, περνάμε στο άνοιγμα διοργανικών διαπραγματεύσεων ε, και τη διαπραγματευτική ομάδα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. δεκτή. 43 υπέρ 6 κατά καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Και έχω τον κατάλογο εδώ της διαπραγματευτικής ομάδας, εάν θέλετε να το δείτε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσω για την ψηφοφορία και να σας συγχαρώ και για την ποιότητα του διαλόγου που είχαμε σε ό,τι αφορά τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Thank you, σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 κατάλογος τρίτων χωρών που οι υπηκοοί τους πρέπει να έχουν θεώρηση για τη έλευση των εξωτερικών συνόρων και κατάλογος των τρίτων χωρών που εξαιρούνται αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής. Ο κ. Δίας Δεμέρα είναι εισηγητής. Έχουμε το σχέδιο έκθεσης ε, πριν πάμε σε διοργανικέ σε διοργανικές διαπραγματεύσεις. Θέλει να πει κάτι ο εισηγητής. Πρέπει να ψηφίσουμε. Μην περνάμε στην ψηφοφορία. Ωραία. Περνάμε στην ψηφοφορία. Και ξεκινάμε. Α, συγγνώμη, στο σημείο 4 έπρεπε να πάμε. Να υπήρχε κι άλλο. αδελφοί, αφού την έκανα τώρα την εισαγωγή, δεν ψηφίζουμε το 6 και πάμε μετά στο ΦΠΑ. Ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση Δίας Δεμέρα. Σας πειράζει? Και θα επανέλθουμε στο 4. Εντάξει όλοι. Αν έχετε πρόβλημα πείτε μου. Συμφωνείτε? Yep, we're ready. My apologies, but we can we'll we'll, we'll proceed with uh, Mr. Diaz de Okay, let. Ε, ε εγώ αυτό λάθος, συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Συμβιβασμός μέρος Α, ο μηχανισμός. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική μέρος Β. Πράξη κατά εξουσιοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 23 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Άρχιε τη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. πέρας δεκτό με 42 ψήφους υπέρ 9 κατά. Και τώρα ψηφίζουμε για την έναξη διαπραγματεύσεων για διαπραγματευτική εντολή και σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών. τη η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. 42 υπέρ, 9 ψήφοι κατά, μία αποχή συγχαρητήρια στον κύριο Δίας Δεμέρα. And now colleagues Και συνάδελφοι, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά πάνω στο σημείο 4. Α, σε ό,τι αφορά τη διαμορφώση ενός ε, οριστικού συστήματος για το ΦΠΑ και την καταναλώνηση της ε, φοροαπάτης. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Χουάν Φερνάντο Λόπος Αγγιλάρα. Πρόκειται για την έγκριση σχεδίου γνωμοδότηση και αν δεν θέλει το λόγο ο εισηγητής μπορούμε να περάσουμε πάρα αυτά στην ψηφοφορία. Τροπολογία 9, συνάδελφοι. Είστε έτοιμοι. Έναξη ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Διοκτώ, λέει ο πρόεδρος. Okay, colleagues, τρία, πρόεδρε, συναδελφοί. Τη δύο την ψηφίσαμε, την ψηφίσαμε τη δύο. Okay, sorry. So colleagues, um, we voted on... Συνάδελφοι, να ψηφίσουμε και την 8, όχι μόνο την 9. Την 8 λοιπόν ψηφίζουμε, ζητώ συγγνώμη. Έναρξη. Την 8. Πέρασε, εγκρίνεται τώρα τη συμβαστική 2. Στη συμβαστική 2 είμαστε και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η ψηφοφορία τώρα ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 15. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Οι 2 στην τελική σκέψη ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ένα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον συγκεκριτή. Στις 13 Ιουλίου ψηφίζει και η Οίκον. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίε. Έχουμε άλλη ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Συνάδελφοι, αν θέλετε να φύγετε, να κάνετε ησυχία παρακαλώ, γιατί έχουμε άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Το 7, που είναι Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό Έτο 2017, η κυρία Μακοβέη είναι η εισηγητριά. Καλέ διακοπέ σε όλου σα, αλλά έχουμε και ένα θέμα ακόμα. εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης και η κυρία Μακοβέη θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης ε, και για το σχέδιο του προπολογισμού για όσους θέλουν να μείνουν. 22 Αυγούστου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογίων, γι' αυτό και το συζητάμε τώρα αναγκαστικά. Σας παρακαλώ, ησυχία στην αδελφή. Και ακριβώς επειδή έχουμε τα προβλήματα αυτά και τα βιαστούμε, κάνουμε την παρουσίαση της έκθεσης τώρα. Make your presentation. Thank you. Mrs. McAvey, you have the floor. Κύριε Μακοβέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, τα πιο σημαντικά σημεία σε ό,τι αφορά τον ε, προπολογισμό της Κομισιόν το 2017 είναι τα εξή. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητοι πόροι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και τα εξωτερικά σύνορα και σε ό,τι αφορά την παροχή υποστήριξη για την υποδοχή ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Κατά δεύτερο, χρειάζεται αλληλεγγύη με όσου βρίσκονται σε καθεστώ πραγματική ανάγκη, καθώ και διατηρεί. Κύριε Μακοβέη, διακόπτει ο Πρόεδρο.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 Sorry, Mrs. just Όπως έλεγα λοιπόν, η γραμματοδότηση αυτή για τη ΛΥΜΠΕ για τον ε, Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για το 2017, όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να δίδονται οι απαραίτητοι πόροι για να προστατευτούν τα εξωτερικά σύνορα, να ενισχυθεί η ασφάλεια και να δοθεί η υποστήριξη που χρειάζεται στα κρατημέλη για την υποδοχή ατόμων που χρήζουν διεθνού βοήθεια. Χρειάζεται αλληλεγγύη και διατήρηση της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών όταν ε, απειλούνται από την τρομοκρατία και από στοιχεία τα οποία διαταράσσουν ε, τις αξίες μας. Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να πετύχει ε, το πολιτεστημοσιονομικό πλαίσιο είναι να μας δώσει τις δυνατότητες να αντιδράσουμε πιο καλά στις ανάγκες του 2017. Απλοποίηση επίσης των ε, δημοσιονομικών κανονισμών και του δημοσιονομικού πλαισίου και κάποιοι τομείς όπως ο τίτλος 4 ε, ε, έχουν μειωθεί εδώ οι δαπάνε λόγω της περιπλοκής του συστήματος. Θα πρέπει όλα αυτά να απλοποιηθούν και εκ παραλλήλου να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πώς πάρουν τα χρήματα τρίτο σημείο. Καλωσορίζω την ε, χρηματοδότηση με 1,6 δις ευρώ του Ταμείου για τους Μετανάστες και το, ιστορικό, ε, το Ταμείο Ιστορικής Ασφάλειας, 0,7 δις, ε, καθώς και τη συνολική χρηματοδότηση για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη Φυλακή και την Αυτοφυλακή. είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει σωστή ανθρωπιστική αρρωγή για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζουν την αύξηση των πόρων για τις ε, υπηρεσίες δικαιοσύνη και ιστορικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και τη σταθεροποίηση και είναι σημαντικό παράλληλα να δικαιολογηθούν ε, οι μεγάλες αυξήσεις ε, στον προπολογισμό του EU LISA πάνω 52%. Ξέρουμε ότι αυτό έχει να κάνει και με την ε, συνθήκη του Λονδίνου, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ε, γίνεται η κατανομή των πόρων μεταξύ ISF και η Γιουλίζα. Οι δαπάνες θα πρέπει να δαπανούνται, να εκχωρούνται ε, ανάλογα με τις προτεραιότητες και θα πρέπει να δούμε και κεφάλαια τίτλους όπου ενδεχομένω χρειάζονται ε, λιγότερες δαπάνες ε, και μόνο μετά θα πρέπει να ζητάμε νέε πόρε. Και τέλος, θα πρέπει να ανταποκριθούμε ταχαίως στις μετατραπόμενε ανάγκε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, επόμενες τις βασικές αξίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Thank you very much. We, um, has anyone asked for the floor? No one has asked for the floor. Uh, Um, Ζητάει κανείς το λόγο, όχι. Ο κύριος Ντεπρέ, α, ο κύριος Δουπρέ και η κυρία Σπινέλη. Ε, Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ντεπρέ, αγαπητοί συνάδελφοι, για να σας πω τις σκέψεις μου είναι τεχνικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι σε σχέση με το πολιετές πλαίσιο μιλάμε για την περίοδο 17-20 και επικεντρωνόμαστε στο 2017 κυρίως όσον αφορά το πολιτές πλαίσιο το οποίο δεν καλύπτει βέβαια μόνο το 17 εξορισμού είναι από το 17 μέχρι το 20 οπότε μιλάμε ότι για τροπολογίες που θα πρέπει να κατεβάσουμε ούτω ώστε να δούμε το πλαίσιο αναφοράς δεν είναι μόνο η επόμενη χρήση αλλά είναι η περίοδος μέχρι το 20 τώρα όσον αφορά την πρώτη παράγραφο εδώ διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι προσέχουμε την ε, διάσταση ασφάλεια. Είναι κορυφαία προτεραιότητα το μεταναστευτικό και η διαχείριση των ροών. Οπότε και εδώ θα κατεβάσω κάποια τροπολογία. Επίσης, όσον με τις διάφορες υπηρεσίες, συμφωνώ ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε για την αύξηση της πληκοδότησης για το ίδιο e Λίζα ε, πάντως πρόκειται για στρατηγικό θέμα. Εμείς ε, το θεωρούμε αυτό προτεραιότητα. Αυτή την παράταση της αποστολής και την πληκοδότηση που είναι απαραίτητη για την υπηρεσία αυτή και για την ΕΑΣΟ, μια που είναι κάτι στρατηγικά σημαντικό για το μέλλον της πολιτικής ε, υποδοχής και το μεταναστευτικό γενικότερα. Αυτά προς το παρόν, Πρόεδρε. Η Μπάρμπαρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για το σχέδιο κειμένου και για την παρουσίασή της και από πλευρά μου έχω να πω ότι σε πολλά σημεία επιδέχεται βελτίωση το κείμενο και θα πρέπει βέβαια να αξιοποιήσουμε τη δουλειά των προηγουμένων ετών και οπότε και εμείς με κάποιες τροπολογίες θέλουμε να χτενίσουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία δηλαδή ο διαχωρισμός σε όλα τα σχέδια προπολογισμού των δαπανών για την ενίσχυση των ε, στρατηγικών της, ε, του επαναπατρισμού ε, και επίσης κάποια έξοδα για την νόμιμη μετανάστευση. Οπότε και αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να προάγουμε την ιδέα μιας αυθεντικής ένταξης. Επίσης να υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για έρευνα και διάσωση ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να υποστηρίξουμε ε, ε, το τι πρέπει να γίνει σε διάφορες χώρες ε, μέλη για να διαχειριστούμε τις ροές. Επίσης συγκεκριμένοι πόροι. Συγκεκριμένη πόρη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια φαινόμενα τα οποία είναι ολοένα και πιο ενισχυτικά όπως η αύξηση του αντισημιτισμού, όπως η Ισλαμοφοβία, η Εφροφοβία, επίσης ο φόβος και το μίσος κατά των τσιγκάνων σε διάφορα κρατη Άρα ε, η σχετική πόροι προς τα τρίτα κράτη δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την θέληση, την ικανότητα των ε, φιλικών μας χωρών να συμμετάσχουν στον έλεγχο της μετανάστευσης. Θα πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες ε, πανυποδοχής. και πρέπει να δούμε το πώς δεν θα φύγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών στην Ευρώπη και των ετούντων άσυλο επίσης και να δούμε το πώς δεν θα νομιμοποιήσουμε ε, δικαιοδοτικά καθεστώτα. Αυτά δεν θα τα εγκρίνουμε εμείς επίσης σε εθνικό επίπεδο να υπάρχουν εγγύσει μηχανισμών για διαφάνεια και έλεγχο όσον αφορά ε, την ευθύνη των διαχειριστών των ευρωπαϊκών πόρων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία, θα πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διαδρομή εποπτεία και όχι μόνο ex post. Ε, οπότε έτσι θεωρούμε ότι πιο εύκολα θα πετύχουμε τους στόχους μας. Τέλος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να περιχαρακώσουμε κάποιο είδους κριτήρια, ποσοτικά και ποιοτικά. Έτσι να μετρήσουμε το αν πιάνουν τόπο τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Τα έγγραφα, οι έκθεσεις που έχουν σχέση με τα κοινοτικά χρήματα νομίζω ότι θα πρέπει να ε, δημοσιοποιούνται κατά τη γνώμη μας. Και ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ κύριο Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Μπόνι. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά. Βλέπω πως θα έχουμε επιπρόσθετες πηγές για την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες που ξέρουμε πως είναι σοβαρό πρόβλημα και έχουμε όλο και περισσότερες ουσίες να αξιολογήσουμε. Από την άλλη έχουμε την μείωση στη ροή εργασίας και κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό για το 2017 έως 2020 σκοπεύουμε να διαθέσουμε να αναθέσουμε στην νέα αυτή υπηρεσία το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης κινδύνου. Είναι σαφές για μένα πως το σχέδιο αυτό για την περίοδο 2017 έως 20 θα πρέπει να περιλάβει περισσότερους πόρους για αυτή την υπηρεσία. Θα κάνω μια σχετική τροπολογία. Σας ευχαριστώ. Η Μόνικα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πω μόνο το εξής. Το πρώτο είναι για τους συζητητές. Είχαμε μια πολύ σοβαρή ακροάση και εκεί πέρα το κέντρο αυτό μας είπε τι συντονισμός απαιτείται μεταξύ των κρατών μελών, ειδικά για την κακοποίηση των παιδιών, την σεξουαλική και μας είπε ότι λόγω έλλειψης προσωπικού δεν υπάρχει συντονισμός. Και αυτό έχει θλιβερές συνέπειες, Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω να είστε σε επαφή με το EC3 για να ξεκαθαρίσετε τα προβλήματα που σχετίζονται με τον προπολογισμό. Να ξεκαθαρίσουμε αν υπάρχει κάποια ανάγκη. Γιατί αυτά τα εγκλήματα εις βάρος παιδιών και μωρών και παιδιών προσφύγων και τα λοιπά πρέπει να παταχθούν. Γιατί έχουν πει ξεκάθαρα ότι δεν είναι σε θέση να δουλέψουν λόγω έλλειψης ε, χρηματοδότησης. Τα ακούσατε όλα για τους ασυνόδευτους αγγλίξους κτλ. Ναι, ναι, το είπα χθε στην Ολομέλεια για τα 10.000 παιδιά. Του ασυνόδευτου ανήλικου που εξαφανίστηκαν. Ναι, ναι, ο Κλοντ ε, το είδε. Έχουμε μια κρόαση ακριβώς για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Την είχαμε μόνο. Και εκεί πέρα η EC3 μας είπε ότι λόγω έλλειψης προσωπικού δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει αυτά τα βαριά εγκλήματα και να συντονιστούν. Και δείτε εδώ πέρα και τα παιδιά των προσφύγων που είναι απροστάτευτα, συνόδευτα, δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν λεφτά κτλ. Ελάτε σε επαφή λοιπόν με το EC3 γιατί μας το είπανε ξεκάθαρα. Και πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά τα εγκλήματα. Και εμείς να επιμείνουμε νομίζω ως Λίμπε. Uh, ναι, εντάξει, συμφωνώ. Δεν είχα ε, κάτι τέτοιο συγκεκριμένο, αλλά επέμενα να υπάρχουν λεφτά για καταστάσεις ανάγκης. Ναι, θα πούμε ότι είναι η προτεραιότητα της ε, ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ να το συζητήσω με τους ε, συναδέλφους μου. Και σας ευχαριστώ για την συμβολή σας. Ναι. Τερέζα, τι έχεις κάτι να πεις. Ναι. Κα, κάτι γρήγορο. μόλις ήρθα θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Χολμαϊρ. Με έχει δίκιο και σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Μακοβέη. Εγώ είχα πάει και μίλησα και με ανθρώπους ε, πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι συνθήκες είναι περίπλοκες ε, για τους ασυνοδευτούς ανηλίκους. Αυτό το οποίο είδα από όλα τα προβλήματα, νομίζω πως το πραγματικό ζήτημα είναι η ασυνοδευτή ανήλικη. Είναι μια ομάδα που ζει σε τρομερές συνθήκες. Υπάρχουν ανήλικοι που είναι με τις οικογένειές τους, έχουν βεβαίως προβλήματα, αλλά ε, από 10 έως 17 ε, οι περισσότεροι είναι σε κέντρα κράτησης, ε, οι περισσότεροι δεν έχουν την ευκαιρία να μετακινούνται. Οπότε πρέπει να τους βοηθήσουμε. Ειδικά αυτή την ομάδα. Για να μην πέσουν στα χέρια διακινητών και να πω πως στηρίζω εδώ πέρα αυτό το οποίο είπε η Μόνικα. Σας ευχαριστώ. Και σας, σας ευχαριστώ για τι συνεισφορά σας στη συζήτηση και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία της τροπολογίες σας. 22 Αυγούστου είναι η προθεσμία και η έγκριση στην Επιτροπή θα γίνει στις 31 Αυγούστου και στην Επιτροπή Budget το Σεπτέμβριο. Θέλετε να πάρετε το λόγο, ναι, Μόνικα και η Τερέζα ήταν τόσο πιστικέ που θα τι καταθέσω εγώ εξ ονόματό μου τι τροπολογίε. Ναι, μα γι' αυτό έχουμε τι συνεδριάσει στην Επιτροπή και γι' αυτό γίνονται και συζητήσει. Ε, Τόμας για το θέμα αυτό Ήθελε να πάρει το λόγο ή για τα διάφορα. Ναι, ήθελα να πάρω το λόγο για τον προπολογισμό. Ναι, συγγνώμη Μόνικα, ήμουν στην Ολομέλεια και είχαν ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον Μπαχρέιν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ξέρετε ότι είναι κατεπήγον το θέμα αυτό και πραγματικά πρέπει να συμμετέχουν. Ναι, ναι, προχωρήστε, λέει ο Πρόεδρο. Για το προπολογισμό του 2017 από πλευρά τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να ταπανίσουμε πιο πολλά χρήματα για τους ε, ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Για μένα το θέμα τη ασφάλεια είναι ουσιώδε. 3 δι ευρώ για την ακτοφυλακή και τη συνοριοφυλακή θέτει ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς θέλουμε και επιθυμούμε να συμμετάσχουμε από πλευράς του ΕΛΚ θα θέλαμε ακόμα πιο πολλά χρήματα σε ό,τι αφορά το 2020 θέλουμε πιο πολλά εργαλεία ευελιξίας και κοιτώντας ε, τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια της ευελιξίας πρέπει να πούμε ότι το 2016 αντιδράσαμε θετικά για την κρίση, για την κρίση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε πιο πολλά χρήματα στον τίτλο 3 και 4. Είναι πολύ βασικά τα θέματα αυτά, θεωρώ. Και έχουμε στο σημείο αυτό τρεις προτεραιότητες. Τρομοκρατία, ριζοστατικοποίηση και Τέτα Τέταρτη προτεραιότητα, τα νέα ναρκωτικά. Τα νέα συνθετικά ναρκωτικά. Και να υποστηρίξω όλες αυτές τις δράσεις. Ναι, το αναφέραμε αυτό. Ανέφερε και η συνάδελφος στις ψυχοτρόπες ουσίες και η βοηθός της κύρια Μακοβέη σημείωσε όλες τις πατρίσει σας. Κάντε λοιπόν τις σχετικές τροπολογίες γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφου και όλο το προσωπικό που ασχολήθηκε με το σημείο αυτό. Θα πάμε στα διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση στις 11 Ιουλίου. Για όσους δεν θα είναι εδώ την άλλη εβδομάδα, Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι. Τους υπόλοιπους θα σας δω στην επόμενη συνεδρίαση στις 3 στις 11 Ιουλίου. Του λέμε την άλλη εβδομάδα.